Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού και ήθελα να επιβεβαιώσω τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίσει ε, στη διαδικασία της Συμφωνίας σύνθεσης της Γεωργίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 10 Νοεμβρίου η Αντιπρόεδρος κυρία Μογκερίνη πήγε στη Γεωργία. Ήταν μια πολύ επιτυχημένη επίσκεψη. Το δεύτερο Συμβούλιο για τη Συμφωνία Σύνδεσης έλαβε χώρα στις 16 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες και ο Επίτροπος Χάν θα είναι στην Τυφλίδα αύριο. Πράγμα το οποίο δείχνει τη δέσμευση σε σε υψηλό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μάλιστα σε εβδομαδιαία βάση. Το Συμβούλιο Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργίας εξέτασε την πρόοδο της εφαρμογής συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ Γεωργίας, η οποία ε, υπογράφτηκε τον Ιούνιο τη περασμένης χρονιάς. Το Συμβούλιο εξέτασε ορισμένες από τι προκλήσει που παραμένουν και ως προς την πρόοδο πρέπει να πω ότι καλωσορίζουμε τη σωστή εφαρμογή ε, της Συμφωνίας Σύνδεσης και της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου ε, Free Trade Agreement και ε, εκεί εξετάσαμε τα θέματα εξαγωγών της Γεωργίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και η προσέγγιση μεταξύ των διαφόρων ε, προτύπων ε, των ΜΕΝ και των ΔΕ προχωρά με καλό ρυθμό και θα πρέπει οι επιχειρήσεις στη Γεωργία να μπορέσουν να δρέψουν τα ωφέλη της Συμφωνίας Σύνδεσης και της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου. Έρχομαι τώρα στις προκλήσεις αγαπητοί συνάδελφοι. Σίγουρα είναι ανάγκη να υπάρξει ένα πολιτικό περιβάλλον, ένα πολιτικό κλίμα με ηρεμία και σεβασμό, βήματα που ε, θα δυναμίτιζαν το κλίμα πρέπει να αποφευχθούν. Σε όλες μας τις επαφές τονίσαμε ότι πρέπει να διατηρηθεί το δημοκρατικό momentum, αυτός ο ρυθμός σε θέματα δημοκρατίας εν ώψη και των ε, εκλογών του 2016 και τονίσαμε σε όλες μας τις επαφές ότι περιμένουμε πλήρη σεβασμό στην ανεξαρτησία όλων των θεσμικών οργάνων συμπεριλαμβανομένων του συνταγματικού δικαστηρίου. Όλων δηλαδή των θεσμών στη χώρα αυτή που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η επικείμενη προεκλογική εκστρατεία θα είναι η πρώτη που θα διενεργηθεί μετά τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Σύνδεσης. Συμφωνούμε με το στόχο ε, διενέργειας ελεύθερων και ήρεμων εκλογών. Αναγνωρίζουμε πλήρως την έκβασή τους ε, ως νόμιμη έκβαση. Η ελευθερία των μέσων μαζικής επικοινωνίας είναι απαραίτητη και αυτό είναι εγγύηση και ε, η επαρκής πρόσβαση των κομμάτων της αντιπολίτευσης στα μίντια είναι ε, προαπαιτούμενο και εγγύηση για να υπάρξει σεβασμός του εκλογικού αποτελέσματος. Και καλωσορίζουμε την ε, βούληση της Γεωργίας να υιοθετήσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης βρίσκεται στο επίκεντρο της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κρίνει επί της ουσίας τις υποθέσεις που φτάνουν στα δικαστήρια. Ασχολείται με το κατά πόσο τηρούνται οι αρχές και αυτό ισχύει και για τις δίκες υψηλού προφίλ όπως αποκαλούνται. Πρόσφατες υποθέσεις όπως είναι οι αγωγές ε, εναντίον του Ρουστάβη του και η... του Ρουστάβη 2, το κανάλι αυτό και ε, η προφυλάκηση των σχετικών ε, στελεχών ε, είναι υποθέσεις που, έχουν, ε, που είναι υψηλού προφίλ. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία ε, της δικαιοσύνης. Το Συμβούλιο Αξιολόγησης της Συμφωνίας Σύνδεσης καλωσόρισε την πρόοδο που έκανε η Γεωργία για την απελευθέρωση των θεωρήσεων το τόνισε αυτό και ο Επίτροπος Χάν και η Αντιπρόεδρος Μογκερίνη. Πολλές, ε, πολλά προαπαιτούμενα έχουν ήδη εκπληρωθεί και θα πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Η τελική απόφαση δεν μπορεί να προβλεφθεί. Βλέπουμε θετικά ε, στοιχεία σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν θετικές εξελίξεις δηλαδή. Τώρα, ως προς τις εξελίξεις της ε, αποσχιστικές περιοχές της Απχαζίας και της Νότιας Οσετίας. Αυτά τα θέματα συζητήθηκαν στο Συμβούλιο Σύνδεσης. Η Αντιπρόεδρος Μογκερίνη και ο Επίτροπος Χάν επιβεβαίωσαν την στεθεναρή τους στήριξη στην εδαφική ακαιρεότητα της Γεωργίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σταθερά προσιλωμένη στην ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων και στην σταθερότητα. Η πολιτική μας για την μη αναγνώριση ε, των, των περιοχών αυτών παραμένει και η συμπροεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των συζητήσεων στη Γενέβη και οι αποστολές παρακολούθησης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα αυτά είναι έμπρακτα δείγματα της δέσμευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συνεργασίας της. Εκφράζουμε την εκτίμησή μας για τη συνεισφορά της γεωργίας στις αποστολές διαχείρισης της κρίσης ε, με ε, επικεφαλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στο Μαλί, στην Ουκρανία και αλλού. Σας, ευχαριστούμε σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και περιμένω ενδιαφέρον να ακούσω τις απόψεις σας για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Ευχαριστώ. Ε, thank Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Επίτροπε. Τώρα οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων θα λάβουν το λόγο. Καταρχήν εξ του ΕΛΚ ο κύριος Στέτινα για δύο λεπτά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αρχίσω ως εξής. Ζήσαμε στη Γεωργία δύο επαναστάσεις του Καντσαχούντε και του Σεβαρνάτζε. Γι' αυτό χαίρομαι γιατί η τελευταία αλλαγή έγινε υπό δημοκρατικές διαδικασίες έτσι ώστε η γεωργία να ε, ξεφορτωθεί το σοβιετικό της παρελθόν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ε, τη δράση του Στάλιν και τα μνημεία που είχαν στηθεί στη μνήμη του. Επίσης, ε, το γεγονός ότι δεν έχουν προσαχθεί πολιτική στη δικαιοσύνη. Δεν πρέπει να, να ξεχάσουμε τη ε, δράση και του κυρίου Σάκασβίλη. Επίσης ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση που αποτελούν βάρος του παρελθόντος και επίσης τον ε, τηλεοπτικό σταθμό ο οποίος διώκεται. Μερικά χρόνια πριν ε, ασχολήθηκα με έναν εγγονό του Στάλιν. Βρίσκεται στην ε, Τυφλίδα. Θεωρούμε ότι δεν είναι επικίνδυνος, αλλά το φάσμα του παρελθόντος υφίσταται και μπορεί να βλάψει τη χώρα. Πέρσι το Δεκέμβριο συνυπογράψαμε μία συμφωνία σύνδεσης, εάν βεβαίως τηρούνται οι δημοκρατικές αρχές και υπάρχει κράτος δικαίου και εξασφαλίζονται οι βασικές ελευθερίες. Εύχομαι να τα καταφέρει η Γεωργία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριος Μποστινάρο έχει το λόγο για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η αναθεώρηση της ε, πολιτικής για την Ανατολική Γειτονία παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα για να ε, και στόχο έχει να δώσει νέα πνοή στις σχέσεις με τις χώρες αυτές. Και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να δώσουμε και μία νέα πνοή στην Ανατολική Γειτονία βασισμένη στην διαφοροποιημένη προσέγγιση ανάλογα με το βαθμό που δείχνουν προς τη μία συνεργασία οι χώρες. Και η γεωργία σε αυτό είναι πρώτη-πρώτη. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη τη σημασία που έχει η γεωργία για μας και θα πρέπει να υποστηρίξουμε μια χώρα και ένα λαό που έχει δείξει σαφή στάση υπέρ της Ευρώπης. Είναι μεγάλο εταίρος η γεωργία στον Εύξηνο Πόντο και αυτό είναι όλο και πιο έντονα στα σημερινά δραματικά με τις σημερινές δραματικές συνθήκες. Έδειξε λοιπόν η Γεωργία την δέσμευσή της με μεγάλη πρόοδο που σημείωσε στις μεταρρυθμίσεις και σε ό,τι αφορά και το σχέδιο δράσης για τις θεωρήσεις. Ελπίζω στο επόμενη, στην επόμενη έκθεση προόδου να επιβεβαιωθούν όλες αυτές οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από τη Γεωργία και προκειμένου να απολαμβάνουν τελικά ένα καθεστώς ελεύθερο από θεωρήσεις οι Γεωργιανοί. Θα πρέπει να πω όμως ότι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε αυτονόητη τη σταθερότητα στη χώρα αυτή. Θα πρέπει να υποστηρίζουμε από πλευρά της Ευρώπης την διαδικασία μεταρρύθμισης, καθώς και την ε, ανεξαρτησία και επικυριαρχία της χώρας, ε, λαμβάνοντας υπόψη και όσα έγιναν το 2008 με τη Ρωσία και τώρα αυτά που έγιναν πρόσφατα με την υπογραφή της ε, συμφωνίας απόσχεσης της Αφχαζίας και της Νότιας Εκ θα πρέπει να διασφαλίσει την σταθερότητα της η Γεωργία με συνεργασία μεταξύ όλων των πολιτικών κομμάτων και τέλος ε, απευθύνω έκκληση προς το ΕΛΚ να σταματήσει επιτέλους να παίζει πολιτικά παιχνίδια στην χώρα της Γεωργίας. Δεν την βοηθάμε, μόνο εχθροί της μπορεί να αποδειχτούμε με τον τρόπο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, αξιότιμε κύριε μπόστεινάρου Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Φώτιγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας οδήγησε σε τεράστιες εντάσεις και σε φόβο στη Γεωργία. και έκανε τη χώρα αυτή να πλησιάσει ακόμα περισσότερο τις δυτικές αμυντικές δομές. Είναι η μόνη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που συμμετέχει στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και έγκαιρης απάντησης. Είναι μια χώρα εξαιρετικά δραστήρια στις προσπάθειές μας για κοινή ε, αμυντική πολιτική. Και αυτό το ανέφερε και ο αξιότιμος κύριος Επίτροπος. Έχει συμβάλει στις δράσεις μας στο Μαλί, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και στην Ουκρανία. Θέλω να ε, συγχαρώ τη χώρα αυτή για τις προσπάθειές της. Ωστόσο, η πολιτική της Γεωργίας δεν είναι τόσο επιτυχημένη παντού, σε όλα τα επίπεδα. Και θα ήθελα να αναφερθώ συγκεκριμένα στην ελευθερία της έκφρασης Είμαι φίλη της χώρας αυτής εδώ και πάρα πολλά χρόνια και υπάρχει πραγματικά πρόβλημα με τον τηλεοπτικό σταθμό Ρουστάβη 2. Είναι πολύ δυστυχές αυτό που συμβαίνει και αρχηγοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκονται στη φυλακή, στη Τυφλίδα και αλλού. Βασίζομαι ε, περιμένω μάλλον να γίνουν αλλαγές στους τομείς αυτούς και στηρίζω την απελευθέρωση των θεωρήσεων για τη χώρα αυτή. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα εκ μέρους του Άλτε ο Χαβιέ Νάρτ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι φίλος της Γεωργίας και του γεωργιανού λαού και γι' αυτό θέλω να μιλήσω με πάσα ειλικρίνη. Όταν το εμπόριο ανακατεύεται με την πολιτική, τελικά γίνεται εμπορική πολιτική και τίποτα άλλο. Και αν δει κανεί τι σημαίνει η υπερπαρουσία των οικονομικών συμφερόντων του κυρίου Ιμπανισβίλη, που είναι το νούμερο 153 στη λίστα Forbes, και εάν δει ε, ποιο, ε, ποια είναι τα δύο τρίτα του ΑΕΠ της Γεωργίας και αν ε, δούμε ότι συνεχώς εμφανίζεται αυτό σε διάφορα κυβερνητικά αξιώματα ότι δηλαδή πρωθυπουργοί, υπουργοί, διάφοροι ηθήνοντες στα βιογραφικά τους είναι πρώην εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις του ελόγου κυρίου, τότε κανείς θλίβεται βαθύτατα γιατί βλέπει ότι μιλούμε για το ίδιο πράγματα, για το εμπόριο και την πολιτική. Δεν υπάρχει ελευθερία και δημοκρατία χωρίς ε, ελεύθερη έκφραση και ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και θα ήθελα να αναφερθώ στην περίπτωση Ρουστάβη 2 του τηλεοπτικού αυτού σταθμού και να πω ότι υπάρχει μια δοκιμασία δοκιμάζεται η αξιοπιστία της χώρας ας, αφήσουμε, ας αφήσουν τη δικαιοσύνη να δράσει, να λειτουργήσει πράγματι η Γεωργία έχει προοδεύσει σημαντικά σε πολλούς τομείς αλλά δεν έχει αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα δεν έχει αποκατασταθεί ε, η ελευθερία του τύπου και θα πρέπει η Γεωργία να εμβαθύνει σε αυτά. Και ας μιλήσουμε και για τους εαυτούς μας. Εάν θέλουμε πραγματικά να διευκολύνουμε την κατάσταση, ε, τότε δεν μπορούμε απλά και μόνο να βγάζουμε δηλώσεις για την ε, Μαύρη Θάλασσα να, δεν μπορούμε να ζητούμε από την Ουκρανία και τη Γεωργία να μπαίνουν στο στρατιωτικό σκέλος και να καλούμε τις χώρες του ΝΑΤΟ να τις στηρίξουν. Είμαστε τρελοί, δεν ξέρουμε πόσο δύσκολα έχει πετύχει το σημείο ισορροπίας στη Γεωργία. Μόνο οι αυτοί μας μας νοιάζουν. Ας είμαστε σόφρονες, ας είμαστε ρεαλιστές. Γιατί ε, το σημαντικό ε, είναι να παραμείνει η ειρηνική χώρα αυτή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα εξ ονόματος Ενωτικής Αριστεράς, ο κύριος Μίλος Λαφ Ράνστοφ, παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε για τη γεωργία που έχει μια υποδομή που έχει πλέον καταστραφεί και η βιομηχανία της έχει καταστραφεί. 11% είναι μόνο του ΑΕΠ στον, στην περιοχή του Καυκάσου. Είναι μια χώρα όμως που έχει σημασία πολύ μεγάλη για τη σταθεροποίηση της περιοχής. Έχει ενεργειακό δυναμικό εξαιρετικό εξάγει και ηλεκτρική ενέργεια που είναι το κύριο αγαθό που εξάγεται πέρα από τα αποστάγματα ίνου και τον ίνο. Είναι επιτέλους η χρονική στιγμή να προσαρμοστούμε σε ένα είδος ε, σχεδίου Μάρσα για την ανάπτυξη της περιοχής του Καυκάσου που θα άνοιγε τον δρόμο, το μονοπάτι για τη συμφιλίωση κατά το παρελθόν στην Γεωργία υπήρχαν πάρα πολλά άτομα, προσωπικότητες Τσοτσαβάλς και Αμπράμς και διάφοροι άλλοι και σήμερα μόνο φτώχεια, δυστυχία και υποβάθμιση βλέπει κανείς. Υπό πολιτιστικού πολιτισμικούς όρους αυτές οι χώρες βρίσκονται πολύ κοντά η μια στην άλλη σε αυτή την περιοχή και έχουν πολύ μεγάλο δυναμικό που θα μπορούσε και θα έπρεπε να αναπτυχθεί. Υπάρχει λοιπόν μια ευκαιρία πραγματικά να αποδειχθεί, να αποδειχθεί ότι η πολιτική μας της γειτονία προς τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης μπορεί να λειτουργήσει θετικά. Δεν είμαστε σε θέση όμως να τη διαχειριστούμε σωστά με τη Μολντόβα, την Μπελαρούς και το ίδιο ίδιο δυστυχώ ισχύει και για την περιοχή του Καυκάσου. Επιτέλου ήρθε η χρονική στιγμή να δράσουμε και να σταματήσουμε μόνο τα κενά λόγια. Και στη συνέχεια ο κύριος Ράνστορφ θα λάβει τον λόγο. Κύριε Ράνστορφ, μια ερώτηση. Δέχεστε μια μπλε κάρτα προς τον κύριο, από τον κύριο Αστροκεβίτσιους. Μάλιστα, φυσικά δέχομαι την μπλε κάρτα, βεβαίως. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ συνάδελφε που είσαστε πρόθυμος να απαντήσετε την ερώτησή μου. Συμφωνώ πρέπει να πω ότι έχει ένα, είναι, μια σημαντική οικονομία θα είχε μεγάλη σημασία για αυτή τη χώρα. Είμαι φίλος της Γεωργίας και εύχομαι κάθε επιτυχία στην Γεωργία. Όμως από τη Σοβιετική εποχή έχουμε 7 ακόμα νέα μνημεία του Στάλιν που ανεγέρθηκαν κατά την τελευταία περίοδο. Είναι ένας εγκληματίας όμως αυτός, ο οποίος έχει διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και μάλιστα ε, σε σχέση με το ότι σκλαβώθηκαν πολίτες ε, στην ε, δική του κυριαρχία. Για αυτά τα μνημεία λοιπόν θα ήθελα μόνο επ' αυτού να υπάρξει τοποθέτηση. Ευχαριστώ. Παρακαλώ έχετε τον λόγο να, απαντώσετε, να απαντήσετε κύριε Ράνστορφ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ερώτηση αυτή βρίσκεται όμως εκτός θέματος που βρίσκεται υπό απόψε. Εγώ δεν είπα καθόλου ότι είναι πολιτικό υπόδειγμα ο Στάλιν ή ο Μπέρια ως προσωπικότητες. Ο Σακασβίλη ήταν εκείνος όπου, που είπε ότι αυτά τα δύο άτομα ήταν ε, παραδείγματα που έπρεπε να ακολουθηθούν. Υπέστη την πίεση του Στάλιν, του σταλινισμού η χώρα μου και αναγκάστηκε να αλλάξει την πορεία της ανάπτυξής της μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό όμως είναι ένα δηλαδή διαφορετικό θέμα είναι ένα θέμα για τους ιστορικούς, για ιστορική συζήτηση και όχι για μας εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Δέχεστε μπλε κάρτα από τον κύριο Πόλτσακ, κύριε. Yes. Ναι, την δέχεστε. Πόλτσακ, Παρακαλώ, έχετε τον λόγο για την ερώτησή σας, κύριε Πόλτσακ. Σας ευχαριστώ πολύ που δέχεστε την μπλε κάρτα με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησα τα όσα είπατε πρέπει να πω και ακούστηκαν θετικά αυτά που είπατε. Όμως αν ζητάτε ένα σχέδιο Marshall να ισχύσει και να λειτουργήσει για τη Γεωργία ή για την ευρύτερη περιοχή του Καυκάσου αυτό δεν θα σήμαινε στη συνέχεια ότι θα μπορούσε η ίδια κατάσταση να δημιουργηθεί όπως τότε που αρνήθηκε εξ ονόματος και για, και για την Τσεχοσλοβακία να υπάρξει πρόγραμμα Marshall. Η κατάσταση γύρω από το σχέδιο Μάρσαλ μετά το 1945 ήταν πολύ πιο περίπλοκη. Η ατμόσφαιρα τότε είχε έντονα ακραία πολιτικοποιηθεί. Το 1947 το 1947 μια πολύ σημαντική ξηρασία έπληξε, περίοδο ξηρασίας την οικονομία της ε, Τσεχοσλοβακίας. Υπήρξε ε, λόγω της ε, ξηρασίας, της λειψιδρίας, έλλειψη τροφίμων και σιτηρών και όλα αυτά επιδίνωσαν την κατάσταση του πολιτισμού όσον αφορά τη σύντησή του. Και η μόνη χώρα που δεν που δεν ζήτησε οποιουσδήποτε όρους ήταν ο Καναδάς. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και τώρα ή για τους πρασίνους η κυρία Χάιντι Χάουταλα παρακαλώ. Έχετε για 1,5 λεπτό τον λόγο. Ε, ευχαριστώ. Παρά όλες τις ελλείψεις και τις προκλήσεις στη Γεωργία, εγώ πιστεύω ότι είναι μια χώρα της Ανατολικής Ευρώπης που δείχνει ότι είναι δεσμευμένη ε, και ενδιαφέρεται για το ευρωπαϊκό της μέλλον και πορεία. Πριν από πέντε χρόνια, εγώ δεν θα πίστευα ότι κάποια μέρα αυτή η χώρα θα μπορούσε να γίνει και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε κατά διάνοια. Ακόμα και τώρα είναι μακριά αυτή η στιγμή, αλλά νομίζω ότι κάνει σημαντική προσπάθεια η χώρα και θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις ευρωπαϊκές της επιλογές, γιατί όπως ξέρουμε η σκιά που ρίχνει η Ρωσία ε, αφορά όχι μόνο τη Γεωργία αλλά κάθε ανατολική χώρα. Σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, πιστεύω ότι οι μεταρρυθμίσεις έχουν συνεχιστεί, έχουν δώσει αποτελέσματα. Επίσης πιστεύω ότι παρά κάποιες ελλείψεις, η μεταρρύθμιση της ε, δικαιοσύνης συνεχίστηκε και φυσικά θα πρέπει να δώσουμε σημασία ε, στις υποθέσεις Ρουστάβη. Ε, για να δείξουμε ότι δίνουμε μεγάλη σημασία στην ελευθεροτυπία και στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης αλλά και της δικαιοσύνης. Έχουμε την ελπίδα και υπάρχουν και τα μηνύματα ότι η συμφωνία δείχνει ότι υπάρχει αρκετή ανεξαρτησία στον τύπο. Εμείς θα πρέπει να προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε και τη Γεωργία και τις άλλες συνδεδεμένες χώρες Ανατολικής Ευρώπης που επιθυμούν να γίνουν ε, μέλος της δικής μας κοινότητας. Ευχαριστώ. Κυρία Χάουταλα. Ο jean Λούκ Schaffhauser για 1,5 λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι. εκπρόσωπε της ε, Επιτρόπου. Εγώ θα μιλήσω λίγο πιο γενικά, πιο γεωπολιτικά αν θέλετε. Περάσαμε από μία στιγμή, από ένα κόσμο με ένα πόλο σε ένα διπολικό κόσμο. Ε, από την ε, την ηγεσία της Αμερικής, τώρα έχουμε δύο πόλους. Ε, για να διατηρήσουν όμως οι Αμερικανοί την ε, ηγεσία τους χρειάζονται την Ευρώπη. Και η Διατλαντική Συμφωνία χρειάζεται την Ευρώπη. Θα πρέπει μάλιστα η Ευρώπη να κοπεί στα δύο. Και να μην υπάρχει πολυπολικό κόσμος και ευρωασιατική συμμαχία. Όλη η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αντίθετα και μιλάει ένας αλθατός εδώ, έτσι. Αυτή η πολιτική που αν ήταν ευρωπαϊκή θα έπρεπε να δημιουργήσει γέφυρες ανάμεσα δύο πολιτισμούς, όπως η γερμανική και η γαλλική, που δημιούργησαν την Ευρώπη, όπως η δυτική με την ανατολική, κυρίως με τη Ρωσία, που θα δημιουργούσε αυτό το, ευρωπαϊκό, το μεγάλο ευρωπαϊκό πολυπολικό σύμπλεγμα, αυτό το αρνείστε. Θέλετε όλες οι χώρες. Σερβία, η Μολδαβία, η Γεωργία, η Ουκρανία να κάνουν μια αποκλειστική επιλογή υπέρ μιας πολιτικής αντίθετης στα συμφέροντα της Ευρώπης. Προδίδετε την Ευρώπη. Θα κριθείτε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουλευτά. Για τους μη εγγεγραμμένους. Ο κύριος Γεώργιος Επιτίδιος. Ευχαριστώ, κύριε η ευρωπαϊκή ένωση θεωρεί τη γεωργία πρωτοπόρο στα πλαίσια της πολιτικής της ανατολικής γειτονίας και στηρίζει την εδαφική της ακεραιότητα και τον τερματισμό των συγκρούσεων στις αποσχιστήσεις επαρχίες της Αμπχαζίας και της Νοτιού Οσετίας. η πολιτική αυτή είναι σωστή πρέπει όμως να εφαρμοστεί και με τον σωστό τρόπο δηλαδή να μην στρέφεται κατά των συμφερόντων της ρωσίας. η ρωσία ήταν και εξακολουθεί να παραμένει ένας σημαντικός στρατηγικός εταίρος για την ευρωπαϊκή ένωση. η πραγματικότητα αυτή έχει φανεί εμφατικά κατά την παρούσα χρονική περίοδο κατά την οποία η συνεργασία με τη ρωσία είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση του isis. συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να εξακολουθήσουμε την μεταξύ μας αντιπαλότητα χρησιμοποιώντας ως όχημα προς αυτήν την κατεύθυνση τη γεωργία. αντιθέτως πρέπει να υπάρξει ένας ειλικρινής διάλογος και συνεργασία με τη ρωσία τώρα μάλιστα που οι διεθνείς εξελίξεις και συγκυρίες διευκολύνουν μια τέτοια προσέγγιση. εάν μάλιστα ενισχύσουμε την προσπάθεια της γεωργίας για δημοκρατισμό και οικονομική ανάπτυξη σίγουρα θα συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας καλύτερης ευρώπης. τέλος πιστεύω ότι τα λάθη τα οποία τα διαχρονικά τα οποία οδήγησαν την ευρώπη στις τραγικές εξελίξεις των παρισίων μας δίνουν ε, ένα μέτρο πραγματιστικής πολιτικής συμπεριφοράς και θα αποφευθούν στο μέλλον. ευχαριστώ. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που υπάρχει και η ευρωπαϊκή σημαία και θα έπρεπε να λυθεί αυτό το παράδειγμα. Η Γεωργία είναι ένα σημαντικό εταίρο. Οι πολίτε τη ε, Γεωργία είναι σημαντικοί ω Ευρωπαίοι επειδή στρέφονται προ την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουν να συνεργαστούν και συνεργάζονται μαζί μα. Θέλουμε να ενταχθούν στο δικό μα σύστημα αξιών και στο δικό μα οικονομικό σύστημα. Έτσι αυξάνεται η γειτονία. Δεν είναι ελεύθερη από όρου και προποθέσει όμω αυτή η πορεία. Αναμένουμε με αξίε ε, και αρχέ αρχές και κράτος δικαίου και πλουραλισμό και δημοκρατία. Αυτές τις προσμονές τις έχουν και οι πολίτες της Γεωργίας. Επίσης μεταρρυθμίσεις. Η πολιτική και τα κόμματα πρέπει περισσότερο προσεκτική να αντιμετωπίζουν αυτά τα θέματα. Δεν είμαι Γεωργιανός, δεν είμαι Ιταλός, όμως μου αρέσει το πάθος στα πολιτικά πράγματα και οι ηγετικές πρωτοβουλίες. Όμως θα είναι λάθος να υπάρχει η στρέβλωση της συνεργασίας σε σχέση με τους, τη συνεργασία μεταξύ των δημοκρατών θα είναι λάθος ε, όταν εξαντλείται η πολιτική σε ρόλους ε, άγωνους και δεν θα είναι σωστό να ισοπεδώνονται τα μέσα ενημέρωσης. Έχουν υψηλές προσδοκίες οι πολίτες της Γεωργίας από την πολιτική να υπάρξει πρόοδος, ανάπτυξη, να αναπτυχθεί η χώρα με ευρωπαϊκό τρόπο, χωρίς ε, κυδαιμονία και ανάμειξη από τον μεγάλο γείτονα Ρωσία. Αυτό θα είναι εφικτό όταν η γεωργιανή πολιτική συνενωθεί και με συνεκτικότητα εργαστεί για ένα κοινό κοινό στόχο, για τους κοινούς αυτούς στόχους. Όταν το δικό μας ευρωπαϊκό όραμα θα γίνει το όραμα, το όνειρο όλων των Γεωργιανών. Ευχαριστώ. Ε, thank you. Mr. I like your... Σας ευχαριστούμε. Μου αρέσει και το χιούμορ σας ε, κατά τα άλλα κύριε Γκάλερ. Στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο ο κύριος Μαμίκινς παρακαλώ. Παρακαλώ κύριε Μαμίκινς έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ συναδελφοι έφετο εφέτος είναι 23η επέτειος ε, των επίσημων διπλωματικών επαφών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γεωργίας. Οι αμοιβέ σχέσεις μας ε, πάντα στόχευαν στο διάλογο και την εταιρική σχέση. Πέρσι είχαμε την υπογραφή της Συμφωνίας και Σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργίας για την εμβάθυνση και των οικονομικών σχέσεων. Βρίσκονται μεταρρυθμίσεις καθοδών ώστε μέσα από αυτό το πλαίσιο να δοθεί μια, ένα κίνητρο για την ανάπτυξη της Γεωργίας. Πρόοδος για την απελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατηρίων. Η Γεωργία προχώρησε στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις ε, περισσότερο από την Ουκρανία και τη Μολδόβα. Όμως ε, ε, οι χώρες αυτές έχουν την χάνουν ε, απαλλαγής θεωρήσεων διαβατηρίων. Πρέπει εδώ να δούμε και το θέμα της καταπολέμησης διαφθοράς και σε σχέση με τον Γενικό Εισαγγελέα την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, του πλησίματος παράνομου χρήματος καθώς επίσης και το νέο προοδευτικό νόμο για, τους, για την ανάμειξη του κράτους σε θέματα εργασιακά. Συνάδελφοι, ως, ε, όπως είπε είπατε εκπρόσωπος πρόσφατα, η χώρα όχι μόνο αναπτύσσει τις δικές της σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι και διαβιβαστής ε, σε αυτή την περιφέρεια των τάσεων και των ρευμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε σχέση με τις πολιτισμικές και πολιτιστικές παραδόσεις, ε, ιδιαίτερα όσον αφορά και την παράδοση της Γεωργιανής Ορθόδοξης Εκκλησίας, αυτή είναι ακριβώς η εικόνα της σημερινής Γεωργίας. Γι' αυτό και ως εισηγητής από πλευράς Κοινοβουλίου για τα θέματα, το ζήτημα της Γεωργίας και για την προώθηση των σχέσεών μας με τη Γεωργία θέλω να τονίσω αν υπάρχει ένας γείτονας με τον οποίο θα μπορούσαμε να είχαμε πολύ πιο στενές σχέσεις αυτός ο γείτονας είναι η δημοκρατία της Γεωργίας. Ευχαριστώ. Ε, ε, Σας ευχαριστώ. Κύριε Καρίμ, έχετε τώρα τον λόγο. Uh, having just led Εκ μέρους του Κοινοβουλίου ήμουνα επικεφαλής της πρώτης συνάντησης αντιπροσωπείας σύνδεσης με Ευρωπαϊκή Ένωσης Γεωργίας. Θα ήθελα λοιπόν καταρχάς να ευχαριστήσω τον Συμπρόεδρο και τους ομολόγους μας στη Γεωργία και όλους τους συναδέλφους που ε, έπαιξαν το ρόλο τους, τις ομάδες, ε, και που παρέστησαν σε, στις συνεδριάσεις των ομάδων αυτών. Ήταν δύσκολη η αποστολή υπό πολλές έννοιες, αλλά νομίζω ότι πετύχαμε ένα πράγμα. Οι σχέσεις μας να ξεπεράσουν τις ε, κομματικές προσαρτήσεις και να φτάσουν σε ένα επίπεδο σχέσεων κοινοβούλιο με κοινοβούλιο. Τα μελλοντικά ψηφίσματα μπορούν να βασιστούν σε αυτά που πετύχαμε ήδη. Ευχαριστώ την Κομισιόν για την έκθεση στην, για την ε, ζώνη ελευθερού εμπορίου, την ε, εκτεταμένη και βαθιά. Ε, το επόμενο θέμα είναι η απελευθέρωση των θεωρήσεων. Για τους Γεωργιανούς είναι το όνειρό τους αυτό στο άμεσο μέλλον. Υπάρχει το θέμα της Ρωσίας ε, που στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα ε, στο λαό της Αυχασίας και Οσετίας ότι θα πρέπει ε, να επενδύσουν στο μέλλον σε αυτό. Φυσικά έχουμε και τις εκλογές που πλησιάζουν πολύ σύντομα και είναι σημαντικό λοιπόν η Γεωργία να δείξει τη δεσμευσή της στις ευρωπαϊκές αξίες. Και αυτό δείχνει, μπορεί να το δείξει καλύτερα με την ελευθεροτυπία με το να εκφράσει και να επιτρέψει στα ΜΜΕ να εκφραστούν ελεύθερα. Ευχαριστώ, κύριε καρίμ. Ο λόγος στο κύριο Μεσερίξ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ για τις εξελίξεις στη Γεωργία. Ελπίζω να είναι δικαιολογημένες οι αξιολογήσεις σας. Η Γεωργία έχει κάνει πάρα πολύ πρόοδο από, από όταν κατέκτησε την ανεξαρτησία της, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Ε, και ε, είχε ε, συνταγματικές αλλαγές ειρηνικές και η αλλαγή κυβέρνησης δεν είναι κάτι και καθεστώτος δεν είναι κάτι το ασήμαντο τούτων λεχθέντων θα πρέπει να πω ότι η πολιτική σταθερότητα δεν είναι ποτέ δεδομένη, δεν είναι κάτι που πρέπει να θεωρείται ε, δεδομένο. Πρέπει συνεχώς να αγωνίζεται κανείς για την πολιτική σταθερότητα και αυτό συνεπάγεται τον σεβασμό της αντιπολίτευσης που είναι εκ των ον ουκ άνεφα για να υπάρχει δημοκρατία. Θα πρέπει όλοι να εργάζονται για αλλαγή δημοκρατική ε, της διακυβέρνησης. Ένα σημείο που θα ήθελα να τονίσω ε, τον Οκτώβριο του 2013 οι δημοσιεύσεις έδειξαν ότι υπάρχει 12% υποστήριξη για προ-ρωσικά κύματα, ε, κόμματα και αυτή είναι ο κίνδυνος που πρέπει να αποφύγουμε. Andrej Penković. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Η Γεωργία είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το πλαίσιο της ανατολικής Γετονίας. Η χώρα αυτή απέδειξε ότι τις αναγκές μεταρρυθμίσεις της υλοποιεί. Κατά τη διάρκεια της, ε, των γεγονότων του 2003 υπήρχε μεγάλη παράδοση της ρωσικής ε, επιρροής ε, σε μια χώρα που όμως βλέπει ότι έχει ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Δυστυχώς πληρώθηκε υψηλό αντίτιμο λόγω της του αποκλεισμού από τη Ρωσία και λόγω του πολέμου στην Απχαζία και στην Οσετία. Η Συμφωνία Εμπορίου θα δώσει κίνητρα για τις περαιτέρω αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Όμως τα πρόσφατα γεγονότα σε σχέση με τα όσα συνέβησαν στην Γεωργία ε, μας ανησυχούν. Επίσης η πίεση όσον αφορά την αντιπολίτευση. Στην αποστολή μας στη Γεωργία είχα συμμετάσχει κι εγώ είδαμε την επιλεκτικότητα από πλευράς δικαιοσύνης και των παρεμβάσεων των δικαστικών σε σχέση με την αντιπολίτευση. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση σε σχέση με το έτος εκλογών. Διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο τα μέσα ενημέρωσης, ο τύπος. Χρειαζόμαστε μια ελεύθερη και σε δίκαιο πλαίσιο διεξαγωγή προεκλογικής εκστρατείας. Ελπίζω ότι θα μπορέσει να δραχθεί της ευκαιρίας η Γεωργία Είχαμε και από πλευρά τη δική μα Επιτροπή και του Υπουργού Δικαιοσύνη και Εσωτερικών και ελπίζουμε ότι οι μεταρρυθμίσει θα γίνουν τμήμα του πολιτικού πολιτισμού και από τη Συμφωνία Σύνδεση και ε, εταιρική σχέση και με τη διευκόλυνση θεωρήσεων διαβατηρίων θα βοηθήσουμε τη Γεωργία να ακολουθήσει την ευρωπαϊκή της πορεία με επιτυχία, μια και είναι σημαντική χώρα για την ανατολική γειτονία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Στην συνέχεια Πύρη. Ευχαριστώ. Η Γεωργία από πολλέ ε, πτυχέ είναι μια επιτυχία. Είναι η μόνη χώρα στην περιοχή που κατάφερε να μεταβεί ειρηνικά από τη μία κυβέρνηση σε άλλη. Ε, δεν υπάρχουν όπλα στους δρόμους, αλλά ο κόσμος πάει στις κάλπες είναι μία από τι χώρε Ανατολική Γειτονία που δήλωσε ότι θέλει στενότερη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Συμφωνία Σύνδεση είναι τα θεμέλια αυτή τη σχέση. Μία σχέση που βασίζεται σε αξίε. Ε, τα ανθρώπινα ε, δικαιώματα, η ελευθεροτυπία και το κράτο δικαίου βρίσκονται στην καρδιά αυτών των αξιών. Είναι σημαντικό ακόμα και η αίσθηση ε, πολιτική εμπλοκή στην δικαιοσύνη και στον τύπο να αποφευθεί. Ε, για να το πω διπλωματικά, ε, η υπόθεση του Ρουστάβη θα έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Αλλά είναι ανησυχητικό επίση που ο, πρώτο, ο πρώην πρόεδρο Σακασφίλη προσπάθησε να χρησιμοποιήσει αυτή την υπόθεση για να δημιουργήσει αναστάτωση. Και δεν είναι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η Γεωργία αυτή τη στιγμή. Η Γεωργία θα πρέπει να κάνει τι μεταρρυθμίσει. Ε, Επίση υπάρχει τόσο πολλή αστάθεια στη χώρα που δεν μπορεί να επιτρέψουν οι να υπάρξουν ε, διαιρέσεις απειλές είναι εξωτερικές. Τρία χρόνια μετά ε, τα προβλήματα θα πρέπει να ενωθούν τώρα οι πολιτικές δυνάμεις. Ε, η συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γεωργίας θα μπορούσε να ε, λάβει συγκεκριμένη μορφή αν καταργηθούν οι θεωρήσεις. Ε, αυτό όμως θα μπορούσε να αμφισβητηθεί αν υπάρχει πολιτική αναστάτωση στην χώρα. Υπάρχουν άλλα πολιτικά προβλήματα στη Γεωργία. Ναι, φυσικά. Κάποια η λογική ότι ο νικητής ε, έχει κάθε δικαίωμα ε, κυριαρχεί. Ε, η αίσθηση ότι ο νικητής δεν λογοδοτεί. Επίσης, προ όλο και αναδύονται ακραία κόμματα. Παρ' όλα αυτά είμαι πεπισμένη ότι αν γίνει σοβαρή προσπάθεια από όλε τι πολιτικέ δυνάμει στη χώρα, οι απαραίτητε μεταρρυθμίσει που έχουν ξεκινήσει υπό την προηγούμενη κυβέρνηση θα συνεχιστούν και οι γεωργιανοί πολίτε γρήγορα θα δρέψουν τα ωφέλη από μια στενότερη Συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργίας. Ευχαριστώ. Η κυρία Κουσλός Καραγεύστο, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να πω ότι μεταξύ όλων των χωρών της Ανατολικής Γειτονίας η Γεωργία αναπτύσσει με ταχύτερο ρυθμό την εξέλιξή της προς την δημοκρατία και τον πλουραλισμό. Έχει βελτιώσει τη βαθμολογία της σε όλες τις επιδόσεις η Γεωργία. Μια θετική διακυβέρνηση και δικαιώματα των πολιτών. Αυτά είναι γεγονότα. Είναι επίσης γεγονός ότι τα μη φιλευρωπαϊκά κόμματα θα μπορούσαν εκεί να υποστούν κάποια επιδείνωση λόγω των αντευρωπαϊκών δυνάμεων που όλο και ενισχύονται και αυτό εξηγείται με τα σφάλματα των κυβερνώντων. Για παράδειγμα είχαμε και ένα σκάνδαλο παρακολουθήσεων και παράνομων παρακολουθήσεων τηλεφώνων και πολιτών. Είδαμε ότι υφίστανται τα ίδια προβλήματα όπως με την περίπτωση Ρουστάβη 2. Κατά τα άλλα και στις περιοχές Απχαζίας και Οσετίας η κατάσταση είναι ε, αναλύωτη, αμετάβλητη και γι' αυτό πρέπει να επιμείνουμε να τηρήσει την ευρωπαϊκή της πορεία η Γεωργία. Θα ήθελα να αναφερθώ στις θεωρήσεις διαβατηρίων. Γίνεται προσπάθεια για τη διευκόλυνση θεωρήσεων διαβατηρίων. Αυτό θα ήταν προς αμοιβαίο όφελος. Υπέρ της Γεωργίας και υπέρ της ΕΕ. Όχι μόνο πολιτικά αλλά και οικονομικά. Η Γεωργία χρειάζεται μεγάλη μεγαλύτερη εμπλοκή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των μέσων και στον τομέα των δημόσιων σχέσεων και ενημέρωση ώστε να μην μπορεί να στέφεται με επιτυχία το εγχείρημα τη Ρωσία να επηρεάσει τα τεκτενόμενα. Πρέπει όμω να διατίθενται πληροφορίε και προ του πολιτικού οι πολιτικοί να μπορούν να αναγνωρίζουν τα ασφάλματά του και να υπάρχουν αντικειμενικά γεγονότα και πολυμορφή απόψεων που πρέπει να είναι διαθέσιμε στου πολίτε. Θέλω να ερωτήσω τον Επίτροπο ποιε πρόοδοι υπάρχουν όσον αφορά τι διευκολύνσει θεωρήσεων διαβατηρίων. Πώ έχει το πράγμα και για την υποστήριξη για τα μέσα επίση για την ελευθερία των μέσων στη Γεωργία. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Και τώρα περνάμε στην διαδικασία Catch the Eye, λέει ο πρόεδρο. Ο κύριο Έντουαρτ Κούκαν έχει πρώτος τον λόγο. Παρακαλώ κύριε Κούκαν. Ευχαριστώ πολύ. Στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας θα ήθελα να διευκρινίσω ότι οι χώρες οι οποίες θέλουν στενότερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηριζονται πλήρως, αλλά θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι αυτές οι χώρες πρέπει να έχουν ορισμένους κανόνες και πρότυπα. Η Γεωργία είναι χώρα που δείχνει αφοσίωση ε, στην Ευρώπη με σύνδεση πολιτική, και για οικονομική ένταξη. Θα πρέπει να την υποστηρίξουμε στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να προστατεύσουμε την εδαφική της ακαιρεότητα. Θα πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη στην ενεργειακή κοινότητα. Επίσης θα ήθελα τους ηγέτες της Γεωργίας να τους ενθαρρύνω να αγωνίζονται ε, στην, ε, στο κοινοβούλιο και όχι να υπάρχουν ε, κρατή, φυλακίσεις προδικαστικές. Ο κύριος Μαριάς παρακαλώ έχει τον λόγο. Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργία είναι ιδιαίτερα σημαντικέ, καθώς η χώρα αυτή αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ασφάλεια της περιοχής του Καυκάσου η γεωργία έχει αναδειχθεί σε πρωτοπόρα δύναμη για την εμπέδωση και τη λειτουργία της ανατολικής σχέσης. η ανατολική σχέση πρέπει κατά κύριο λόγο να αποσκοπεί στην ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων της ευρωπαϊκής ένωσης με τα αντίστοιχα κράτη και βεβαίως με τη γεωργία. πρέπει να αποσκοπεί στη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της ένωσης στη διαμόρφωση σχέσεων στη βάση του αμοιβαίου ωφέλους στην ενίσχυση του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών όμως η ανατολική σχέση δεν θα πρέπει να αξιοποιείται από ορισμένες πλευρές ως ένα μέσο επέμβασης στην εσωτερική πολιτική ζωή της γεωργίας. η γεωργία πρέπει να αφαιθεί ανεπηρέαστη να καθορίσει κυρίαρχα την εσωτερική της πολιτική ζωή μεριμνώντας ταυτόχρονα για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της δημοκρατίας των πολιτικών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. μόνο με αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί να εξελιχθεί θετικά η πολιτική κατάσταση στη γεωργία εν ώψη των εκλογών που θα γίνουν το 2016 για τη διενέργεια των οποίων πρέπει να διασφαλιστεί η πολυφωνία και τα δικαιώματα της αντιπολίτευσης. ευχαριστώ. ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μαριά. Και τώρα παρακαλώ. Κιουτσούκ. Έχετε τον λόγο κύριε Κιουτσούκ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, η Γεωργία είναι μια χώρα με πλούσια ιστορία και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αποτελεί μέρος τμήμα της ευρωπαϊκής ιστορίας και πριν από ένα έτος είχε ερτάστηκε η επέτειος της υπογραφής της Συμφωνίας Σύνδεσης. Συντριπτικό ε, ποσοστό του πληθυσμού υποστήριξε αυτή τη συμφωνία καθώς και την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ για πολλά χρόνια αποτελούσε τμήμα της Σοβιετικής Ένωσης η Γεωργία και τώρα αναζητεί την ευρωπαϊκή της ταυτότητα ω Ως ε, κάποιος, ε, ως πολίτης από πρώην χώρα σοβιετικής επιρροής αναγνωρίζω το, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Γεωργία για την δημοκρατική της μετεξέλιξη και δεν μπορούμε να ανεχθούμε αναμίξεις. Πρέπει να επιμείνουμε και να εμείνουμε όλοι να σέβονται το κράτος δικαίου την δημοκρατία και την ελευθερία των μέσων. Χρειάζεται την υποστήριξή μας διαρκώς ε, η Γεωργία για να συνεχίσει αυτή την πορεία της. Ε, ε, ευχαριστώ. Ο κύριος Σόλτας θα λάβει τώρα τον λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ακούσαμε πολλά θετικά σχόλια, καλά λόγια για την Γεωργία απόψε. Ωστόσο, παραμένει το ερώτημα τι είναι ρεαλιστικό τούτων δεδομένων. Τα στοιχεία, τα όσα έχουμε στη διάθεσή μας, οι πληροφορίες που έχουμε είναι σημαντικά και σημαντικές. Πώς θα αναφερθούμε και πώς θα αξιολογήσουμε αυτή την πρόοδο. Πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα κριτήρια. Γι' αυτό ζήτησα να παρέμβω. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεργαστούν με το Συμβούλιο της Ευρώπης το Συμβούλιο της Ευρώπης διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την αξιολόγηση των θεμάτων των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δικαιοσύνης, της ε, ελευθερίας των μέσων του τύπου. Θεωρώ, πιστεύω ότι είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης να συνεργαστούν στενότερα σε αυτούς τους τομείς, διότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει ήδη θέσει υψηλά τον πύχη για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σόλτες. Ε, ο τελευταίος ομιλητής. Πρόεδρε, το 2012 έγιναν εκλογές και κέρδισε ο Σακασφίλη. Ήταν δημοκρατικές οι εκλογές. Η Γεωργία έκανε μεγάλη προσπάθεια στα πλαίσια της μετάβασης. Η χώρα έχει μεγάλο ενεργειακό δυναμικό, αλλά είναι βασικός σύμμαχος της Ευρώπης στον Κάφκασο. Γι' αυτό καλωσορίζω τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν σε αυτή τη χώρα και θα πρέπει να συνεχιστούν απαρασάλευτα αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Και θα πρέπει να σταματήσουν οι πολιτικές ε, πιέσεις και εντάσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πόλτσακ. Ο κύριος Τηλιανίδης, από την Επιτροπή. Thank you, President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπα στην εισαγωγική μου ομιλία, παρακολουθούμε στενά εάν οι κοινέ μας αρχές είναι σεβαστές και βεβαίως αυτό το πράττουμε ως εταίροι μαζί με την Γεωργία. Όντας πεπισμένοι ότι η ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλιστεί διαφανής, ευήμερη γεωργία που είναι προς το κοινό μας συμφέρον. Όλα αυτά συνάδουν με τις προτεραιότητες που ορίστηκαν ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων η ε, Φεντερίκα Μογκερίνη ενθαρρύνθηκε από τον επικοδομητικό τόνο της ε, κυβέρνησης και τους πολιτικούς ηγέτες στην Γεωργία και την αντιπολίτευση που αναγνωρίζουν την ανάγκη να ε, διατηρηθεί η προτεραιότητα για τις μεταρρυθμίσεις και να δημιουργηθεί ένας χώρος ασφαλής ούτως ώστε να προετοιμαστούν καλά οι βουλευτικές εκλογές του επομένου έτους. Σχετικά με την απελευθέρωση ε, σχετικά με την απελευθέρωση των θεωρήσεων βασίζεται στο αποτέλεσμα της αξιολόγησης που έγινε τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, βάσει των πληροφοριών που έδωσαν οι αρχές της Γεωργίας και εμείς θα κάνουμε το Δεκέμβριο μια αναφορά σχετικά με την κατάσταση. Όταν θα έχουμε μια τελική έκθεση, η Κομισιόν θα είναι σε θέση να παρουσιάσει μια νομοθετική πρόταση ούτως ώστε να απαλλαγούν οι Γεωργιανοί από την υποχρέωση των θεωρήσεων και βεβαίως θα είναι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα αποφασίσουν και ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την απόφαση σχετικά με μια τέτοια πρόταση είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Θα ήθελα να κλείσω και πάλι λέγοντας ότι η συμφωνία σύνδεσης με την Γεωργία είναι ένα συγκεκριμένος τρόπος ενεργοποίησης των δυνατοτήτων των σχέσεών μας η εστίαση είναι πάνω στην υποστήριξη, υποστήριξη για βασικές μεταρρυθμίσεις για την οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη, διακυβέρνηση, τομεακή συνεργασία για τις μεταφορές, την ενέργεια και το περιβάλλον. Και βεβαίως όλοι μας έχουμε ε, αισιόδοξη άποψη, διότι Είμαστε ως πολιτική αισιόδοξοι και αυτό πιστεύουμε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ ε, τον